Anatolii Ion că mai pune să mai zică la Stănescu sau doar pentru la agricultură, unde nu am fost de șase luni în 2000. Bonjour. Καλημέρα σας. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλές διακοπές, να είστε ξεκούραστοι, χαλαροί και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το πρόγραμμα εργασιών, το οποίο είναι αρκετά φορτωμένο. Μπορούμε να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις και ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν εγκεκριμένο ως έχει. Πιστεύω ότι είδατε ότι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών συνέβησαν διάφορα στην Ευρώπη, όπως παραδείγματος χάρη πυρκαγιές, καταστροφικές πυρκαγιές στις ε, Μεγάλες Κανάρις νήσους και θέλω να σας πω ότι εξ ονόματος της Επιτροπής έχω στείλει στον πρόεδρο της Περιφερειακής Κυβέρνησης ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Και ανακοίνωσα επίσης ότι είμαστε στο πλευρό της κυβέρνησης ε, των Κανάριων Νήσων αλλά και της Ισπανίας για να συνδράμουμε. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας στο Στρασβούργο συναντηθήκαμε η συνδιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συνεδρίασε και κατά τη διάρκεια αυτής της ε, συνεδρίασης πήραμε την απόφαση το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου της ε, Επιτρόπου Κρέτου θα ανατεθεί στον Επίτροπο Χάν. Πιστεύω ότι θα είδατε ότι έχουν δοθεί τα ονόματα δύο νέων επιτρόπων, μία προσωρινή για την Εστονία, η κυρία Κάνταρη Σίμψον, και επίσης αντικατάσταση της κυρίας Κρέτου ο Ιωάνν Μίρσια Πάσκου. Πήραμε την απόφαση να μην περάσουν από ακρός οι δύο αυτοί οι προσωρινοί επίτροποι, καθότι δεν έχουν αναλάβει το θέμα της συνοχής. Το θέμα της συνοχής, επαναλαμβάνω, το έχει αναλάβει ο Επίτροπος Χάν, τον οποίο συνάντησα πριν τις ε, διακοπές. Αυτά είχα να ανακοινώσω. Και τώρα βεβαίως θα περάσουμε στο θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ σύντομα, δηλαδή την ακρόαση των επιτρόπων όταν ε, αυτοί διοριστούν. Η πρόεδρος Βάντερ Λάιεν και οι επίτροποι που θα αναλάβουν την 1η Νοεμβρίου όπως ξέρετε θα ακολουθήσει ψήφος από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε και προηγουμένως θα υπάρξουν οι ακροάσεις. Εμείς σαν Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων θα ακούσουμε την αρμόδια Επίτροπο για τα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να επεξεργαστούμε το πρόγραμμα των εργασιών και θα υπάρξει σε λίγο η συνάντηση των συντονιστών κατά την οποία θα συζητήσουμε την ε, διαδικασία αυτής της ακρόασης. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία της ακρόασης. Πρέπει να τεθούν όλες οι ερωτήσεις και πρέπει όσο μπορούμε να αποσπάσουμε απαντήσεις. Η ακρόαση αυτή έχει μέγιστη διάρκεια τρεις ώρες και θα λάβει χώρα από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, οι εβδομάδες 40 και 41 δηλαδή. Κατόπιν θα πάρουμε την απόφαση εάν ναι ή όχι δεχόμαστε την υποψηφιότητα του ή Επιτρόπου. Εν ανάγκη μπορεί να υπάρξει και μια δεύτερη ακρόαση διάρκειας ε, μια μισή ώρας, εάν αυτό φανεί απαραίτητο. Τον Οκτώβριο, τη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου στο Στρασβούργο, θα γίνει η ψηφοφορία για την αποδοχή των επιτρόπων. Αυτή είναι η διαδικασία. Μετά την συνάντηση των συντονιστών θα σας παρουσιάσω με ακρίβεια ποια διαδικασία αποφασίσαμε να επιλέξουμε. Για τα μέλη που ήταν ε, μέλη και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου, η ακρόαση της Επιτρόπου Κρέτου έγινε κατά τη διάρκεια της οποίας έθεσαν ερωτήσεις οι συντονιστές και οι απαντήσεις δόθηκαν on block από την Επίτροπο. Πιστεύω και μάλιστα αυτό θα προτείνω στους συντονιστές, ίσως να ήταν καλύτερα να γίνουν οι ερωτήσεις και να δοθούν οι απαντήσεις από τον ή την υποψήφια επίτροπο αμέσως. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια πιο δυναμική συζήτηση και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποσπάσουμε περισσότερες απαντήσεις και πιο ακριβείς απαντήσεις από τον υποψήφιο επίτροπο. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο αυθόρμητη η ερώτηση και η απάντηση σε σχέση με τις ερωταπαντήσεις που προετοιμάζονται από τα μέλη της Επιτροπής είμαστε η συναρμόδια αρχή για την νομοθεσία και θα πρέπει να αναλάβουμε πλήρως το ρόλο αυτό. Αυτά είχα να σας ανακοινώσω και νομίζω ότι μπορούμε αμέσως να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 20. Κατά τη διάρκεια τις συνάντηση που είχαμε στις 23 Ιουλίου, αν θυμάστε, με είχατε διορίσει εισηγητή για τη γνωμοδότηση όσον αφορά την διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2020. Μάλιστα, έχω αναλάβει και την υποβολή των τροπολογιών προς την Επιτροπή Προϋπολογισμού έτσι ώστε να ανασταλούν όλες οι περικοπές που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο και σύμφωνα με αυτά που είχαμε αποφασίσει στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, τον Αύγουστο υπέβαλα αυτές τις τροπολογίες με όλες τις προτάσεις για τα πιλωτικά προγράμματα και τις δράσεις προετοιμασίας οι οποίες είχαν αξιολογηθεί από την Επιτροπή. Πιστεύω ότι είδατε ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμού ήδη έχει εξετάσει αυτά τα πιλωτικά προγράμματα και τα έχει σχολιάσει. Σήμερα σας παρουσιάζω το σχέδιο γνωμοδότησης βάσει της πρότασης της ε, Επιτροπής Προϋπολογισμού για τον προϋπολογισμό του 2020. Το έγγραφο αυτό το έχετε, φαντάζομαι, εξετάσει. Η πολιτική συνοχή είναι μία από τις βασικές αρχές, ένα από τα βασικά εργαλεία που επιτρέπουν να ανταποκριθούμε στις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2020. Και βεβαίως εδώ χαιρετίζω το γεγονός ότι οι πληρωμές αυτές που αφορούν το 2007-2013 πληρωμές συνοχής έχουν εξαντληθεί για την περίοδο 14-20 όλα φαίνεται ότι λειτουργούν όπως πρέπει σύμφωνα με τους προκαθαρισμένους ρυθμούς. Και θα ήθελα να πω για τα νέα μέλη ότι στην προηγούμενη θητεία αντιμετωπίσαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα της κρίσης πληρωμών και μάλιστα πολλές ε, δράσεις δεσμεύτηκαν με αποτέλεσμα να δραστηριοποιηθεί η Επιτροπή μας έτσι ώστε να ρυθμιστεί το θέμα αυτό όσον αφορά την κρίση πληρωμών, η οποία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναληφθεί. Όλες οι περιφέρειες θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να μην βρεθούμε μπροστά σε παρόμοια προβλήματα στην επόμενη θητεία. Στην πρόταση την οποία σας έστειλα ζητώ από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τους την προηγούμενη θητεία, την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αυτά που συνέβησαν έτσι ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε κρίση όσον αφορά το συζύγιο πληρωμών. Πιστεύω ότι ο επαναπρογραμματισμός που αφορά την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων παν, η οποία είχε προγραμματιστεί στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Προτείνω λοιπόν προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών στις 5 την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου Δηλαδή μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου μπορείτε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 2 και 3 Οκτωβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με την διαδικασία, τη συνήθη διαδικασία, θα δώσουμε αμέσως το λόγο στους κοιόδης συζητητές, ξεκινώντας από το ΕΛΚ, την Μαρία Σπυράκη. Μαρία, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που είναι ο προπολογισμό. Και φυσικά θα συμφωνήσω μαζί σας ε, για το θέμα των ε, καθυστερημένων πληρωμών και των σωρευμένων πληρωμών. Έχουμε χάσει αρκετό χρόνο με αυτό και θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ε, κάποιες εξαιρέσεις από τις περιφέρειες δεν είναι αποδεκτές και θα πρέπει να απορροφούνται τα κονδύλια, να εκταμιεύονται εγκαίρως τα διαθέσιμα κονδύλια. Και γι' αυτό θα ήθελα να καταθέσω τροπολογία για την προσθετικότητα. Μόνο έτσι μπορούμε να απορροφήσουμε κονδύλια, όχι μόνο από το PDLTP, αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και πρώτα απ' όλα τις κλιματικές αλλαγές. Και γι' αυτό θα καταθέσω μια τροπολογία με θέμα την σύσταση ενός νέου ταμείου, του Ταμείου της Δίκαιης Μετάβασης, που ήδη έχει εγκριθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και η πρόταση αυτή ε, ήταν πρόταση του καθηγητού Μπούζεκ, του προηγούμενου δηλαδή Προέδρου της Επιτροπής Ήτρε. Και γι' αυτό θα καταθέσω μια σχετική τροπολογία για το Ταμείο της δίκης Μετάβασης. Αυτό το Ταμείο δεν θα είναι μόνο ένα χρηματοδοτικό μέσο, αλλά θα διευκολύνει το μετασχηματισμό της οικονομίας 41 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διευκολύνει επίσης ε, την ανακλιμάκωση και την ανακύκλωση των εργαζομένων, την ε, ανανέωση των δεξιοτήτων του και θα έχουμε πλέον κονδύλια που θα μας διευκολύνουν ε, να εφαρμόσουμε την πολιτική συνοχή στις περιφέρειές μας. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω και από τα άλλα πολιτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την έκθεση μου. Ευχαριστώ και την ε, τροπολογία μου. Ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια για το έργο σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τον Νίνο Πίτσουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που αναλάβατε τη γνωμοδότηση αυτή που αντικατοπτρίζει θαυμάσια θεωρώ τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. στηρίζω και εκτιμώ την προτεραιότητα που δίνεται ε, στην πολιτική συνοχή και τη σημασία του άρθρου 174, δηλαδή να μην αφήσουμε πίσω ουραγό καμία περιφέρεια. Και συμφωνώ και με τις άλλες παρατηρήσεις Και μια και θα είναι η τελευταία χρονιά της τρέχουσας χρηματοδοτικής περίοδου, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επαρκή κονδύλια για όλα τα προεβλεπόμενα προγράμματα, με τις απαραίτητες προσαρμογές φυσικά όπου, είναι, όπου χρειάζονται. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να δώσουμε έμφαση στην περιβαλλοντική κλιματική διάσταση και τους ε, στόχους για την ενέργεια. Σε ό,τι αφορά το 20% δαπάνε για το κλίμα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών για την υλοποίηση αυτού του ποσοστού, αλλά θα πρέπει να εμείνουμε σε αυτό και να το επισημάνουμε. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων εννοείται ότι αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μα και χαίρομαι που φαίνεται αυτό και στην γνωμοδότησή μα που συντάξατε εσείς. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε, κύριε συντάκτη της γνωμοδότησης και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία. Σας ευχαριστώ κύριε Πίτσουλα εκ μέρους της ομάδας Σερινιού ο Όντζε Κνότεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το έργο σας και για την πολύ ισορροπημένη και άρτια γνωμοδότηση που καταρτήσατε. Ελάχιστε θα είναι οι τροπολογίες ε, που θα καταθέσουμε, κυρίως ε, για το κλίμα και τις κλιματικές αλλαγές, γιατί μερικές περιφέρειες ε, έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα από τις κλιματικές αλλαγές και χρήζουν τη δικής μας υποστήριξης και αλληλεγγύης. Χαίρομαι που υιοθετήσατε ισορροπημένη προσέγγιση για να αποφύγουμε την κρίση πληρωμών που είχαμε στο παρελθόν και να μειώσουμε τη... το κενό που υπάρχει μεταξύ ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κνώτεκ. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα, η κυρία Αλεξάνδρα Γκίζε. Σας ευχαριστώ. Εγώ ως μέλος των Πρασίνων φυσικά και θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και την προλαλήσασα που τόνισαν την ανάγκη καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ε, τηρούμε τους στόχους μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 21%, αλλά πώς ε, με αυτό το 21% θα υλοποιήσουμε το συνολικό στόχο του 20%. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις περιβαλλοντικές κλιματικές δαπάνες. Και 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν γι' αυτό. Ε, η ΡΕΚΙ προβλέπει περίπου 30% αυτό του ποσού. Θα χρειαστεί να καταβάλουμε πολύ σοβαρέ προσπάθειε λοιπόν για να υλοποιήσουμε του κλιματικού μα στόχου. Αυτή είναι η πρώτη μα προτεραιότητα και χαίρομαι που τη συμμερίζονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πόσο σημαντική είναι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο τη Δίκαιη Μετάβαση, φυσικά και η πράσινη είναι υπέρ οποιασδήποτε ενέργειας και πρωτοβουλίας που θα διευκολύνει την δίκη μετάβαση και των περιφερειών που εξαρτώνται από τα ανθρακοριχεία και τα χρυσή άνθρακα. Αλλά περιμένουμε την τρομολογία για να δούμε το ακριβές τη περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Η ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας δεν έχει ορίσει ακόμη ισχυώδη Ο Ραφαέλ Φιτό είναι ο του ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησης μπορεί να μας βρει σύμφωνους. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Απλώς τρεις παρακλήσεις, ε, ώστε να αλλάξει το κείμενο και να ενισχύσουμε τρία σημεία, για τα οποία θα υποβάλουμε και τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα για τον τομέα της ανταγωνιστικής οικονομίας και την υποστήριξη των νέων. Έχουν προβλεφθεί 83 δις ευρώ καλό θα ήταν τα κονδύλια αυτά να επαναπρογραμματιστούν για την στήριξη των διευθυντικών υποδομών. Για να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε καλύτερα και το περιβάλλον. Δεύτερο σημείο για την ενίσχυση της άμυνας. 1,5% παραπάνω σε σχέση με πέρσι, σημαντική αύξηση. Κατά τη δική μου την άποψη, θα μπορούσε να υπάρξει υποστήριξη για τα μέτρα των κρατών μελών που ασχολούνται ε, στην μπροστοφυλακή με την καταπολέμηση της μεταναστευτικής κρίσης. Και τρίτον, κλιματικές αλλαγές. Μεγαλύτερη πρικοδότηση και ενίσχυση των κοντιλίων, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είναι απαραίτητη. Και καλό θα ήταν να έχουμε περισσότερους πόρους για τα κράτη-μέλη που πρέπει να αντιμετωπίσουν φυσικές καταστροφές, απρόβλεπτες και πλήττονται από ειδικά φαινόμενα και να αναφερθώ εδώ και στην περίπτωση της ξυλέλα φαστιντιόζα που έχει πλήξει πολλές περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Υπάρχουν και τέτοια προβλήματα επιδημιών ε, που πλήττουν τα φυτά. Θα πρέπει και εκεί να προβλέψουμε την κατάλληλη ενίσχυση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ ο κ. Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δουλειά που έχετε κάνει και μας παρουσιάσατε. Σημερίζομαι πολλές από τις παρατηρήσεις των σκιωδών εισηγητών των άλλων πολιτικών ομάδων που προηγήθηκαν ε, καταθέτοντας επισημάνσεις και προτάσεις. Ε, θεωρούμε αναγκαίο να ενισχυθούν οι προβλέψεις ε, σε κονδύλια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για την νεολαία, ε, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο Ταμείο Μετάβασης, όπως υπόθηκε για να έχουμε μια ομαλή μετάβαση σε μια πιο καθαρή χρήση ενέργειας και γενικά Πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε ως Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, όπως κάναμε και στην προηγούμενη θητεία, τον ε, αγώνα που δίνουμε για να μην αποδυναμωθούν οι πολιτικές συνοχής, κοινωνικής και περιφερειακής. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι το, το κεντρικό ζήτημα όταν συζητούμε τον προϋπολογισμό και τους στόχους της συνοχής. Η πολιτική μου ομάδα θα καταθέσει τις επόμενες μέρες τροπολογίες και φιλοδοξούμε να μην αποδυναμωθεί το σχέδιο που μας παρουσιάσατε, αλλά αντιθέτως να ενισχυθεί υπερασπίζοντα τις πολιτικές συνοχής. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ. Και δύο άλλοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο από την Ομίγυρη. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω διάφορες ιδέες μου. Εγώ δεν έμεινα και πολύ ικανοποιημένος με τη γνωμοδότηση. Μάλλον είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τη γνωμοδότηση και θα ήθελα να σας συγχαρώ. Αν και δεν ήσταν και πολύ επικριτικό σε αυτή τη γνωμοδότηση. Είπατε ότι δεν έχουμε καθυστερήσεις στην προηγούμενη περίοδο 2014-2020 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2007-2014. Ίσως όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας δώσει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις για το θέμα αυτό. Από ό,τι ξέρω, μέχρι στιγμής έχουμε εκταμιεύσει 50% των κονδυλίων της συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 του τέστην το μεγαλύτερο τμήμα της δουλειάς, ο μεγαλύτερος όγκος της δουλειάς θα μείνει για το τέλος της περίοδου. Μιλώ για συν δύο συν τρία χρόνια. Η νέα περίοδος προγραμματισμού θα ξεκινήσει το 2021. Θα έχουμε όμως ακόμη ε, κονδύλια που έχουν μείνει αναξιοποιητά από την προηγούμενη περίοδο μέχρι το 2023. Δεν είναι καλό δεν είναι σωστό αυτό να μεταφέρουμε κονδύλια από τις προηγούμενες περίοδους προγραμματισμού, θα πρέπει να φροντίζουμε τουλάχιστον το ποσοστό απορρόφησης μας θα φτάσει μέχρι 80% τουλάχιστον από την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού και να μην μεταφέρουμε ε, μεγάλο τμήμα των κονδύλιων στην επόμενη περίοδο. Θα πρέπει λοιπόν ε, φέτος και του χρόνου να εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά για να αυξήσουμε το ποσοστό απορρόφησης από την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού για να μην χρειαστεί να τα μεταφέρουμε ενώ θα έχει ξεκινήσει η επόμενη. Όντως, το τελευταίο καλοκαίρι ακούσαμε πολλές ιδέες για τις κλιματικές αλλαγές. Όλοι πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρό είναι το πρόγραμμα, το πρόβλημα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να καταρτήσουμε σοβαρά προγράμματα για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να περάσουμε και στην εφαρμογή. Δεν χρειάζεται μόνο να μιλάμε απλώς για το 20% ή αντίστοιχα ποσοστά θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού, του πυρηνικού εργοστασίου της Ιγναλίνα. Θα πρέπει να παραπληστεί, να κλείσει αυτό το εργοστάσιο. Φαίνεται ότι συνεχίζονται απρόσκοπτα οι εργασίες ε, για το παροπλισμό του εργοστασίου, για το κλείσιμο, ω προ τα τεχνικά σημεία, αλλά υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους τοπικούς πληθυσμούς και για, για το περιβάλλον, για το φυσικό περιβάλλον της Ιγναλίνα. Ε, Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει εκπονήσει καμία μελέτη επιπτώσεων για το θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποια ε, σχέδια μέσα σε ε, ε δύο χρόνια να ε, διαλυθεί ο πυρηνικός αντιδραστήρας, αλλά δεν έχουν γίνει άρτιες ε, τεχνικές μελέτες επιπτώσεων αυτή τη προσπάθεια. Θα πρέπει επιτέλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει κάποιε μελέτε και έρευνε για να εκτιμήσει τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού στου τοπικού πληθυσμού αλλά και στη χλωρίδα και πανίδα και το φυσικό περιβάλλον τη περιοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολλά πυρηνικά εργοστάσια θα κλείσουν στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφή ενημέρωση για την κατάσταση, γιατί στην συνέχεια θα εφαρμόσουμε παρόμοιε πρακτικέ και σε άλλε χώρε. σω θα χρειαστούμε κάποια μέτρα, για παράδειγμα, να, για να αποτρέψουμε την μετάδοση τη ακτινοβολία ή άλλα αρνητικά φαινόμενα. Και ο συνάδελφο Μπούντα ζήτησε το λόγο και τον λαμβάνει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για την γνωμοδότηση που καταρτήσατε και να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις, σύντομες παρατηρήσεις. Στο σημείο 6 καταρχάς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στην ανάγκη μείωση της γραφειοκρατίας για να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Γιατί μία από τις αιτήσεις καθυστέρησης πληρωμών είναι η υπερβολική γραφειοκρατία Επίσης, ε, είναι σαφές ότι στη γνωμοδότηση θα πρέπει να διατρανώσουμε την ανάγκη να μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος, να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να μεταδώσουμε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας η απασχόληση των νέων και σχετική πρωτοβουλία. Επίσης, να αναφερθούμε σε σωστούς ε, μισθούς, ε, δίκαιες αμοιβέ και για την απασχόληση των νέων. Βέβαια, δεν είναι μόνο η απασχόληση πρόβλημα για τους νέους. Το θέμα είναι να έχουν και ε, αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς απολαβές για να μπορούν να ζήσουν, να διάγουν ένα αξιοπρεπή βίο. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για την απασχόληση, αλλά για την ποιοτική απασχόληση για κατάλληλε αμοιβέ. Επίση, ε, οι κλιματικέ αλλαγέ. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε μπροστά στην πραγματικότητα αυτή των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Για να αντιμετωπίσουμε όμω αποτελεσματικά τι κλιματικέ αλλαγέ, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα της βιώσιμης γεωργίας, της αηφόρου γεωργίας. Δεν μπορούμε ε, όμως ε, να αποσυνδέσουμε τα δύο θέματα. Θα πρέπει να συνδυάσουμε την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών με την αηφόρο γεωργία για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τους γεωργούς και να τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν τις γεωργικές τους ε, δραστηριότητες με θετικό όμως αντίκτυπο στις περιβαλλοντικές αλλαγές και κλιματικές αλλαγές. Σας ευχαριστούμε κυρία Βούντα. Η Ρόζα ζήτησε το λόγο ή όχι. Η κυρία Ντονάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να σας συγχαρώ για την γνωμοδότηση. Συμμερίζομαι και το πνεύμα και τα σημεία που σχολιάστηκαν Και επειδή είμαι σκιώδης εισηγήτρια εδώ, ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει για την Ιταλία και ιδίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές όπως η νήσι της Αρδενίας και της Σικελίας, τη σημασία που έχει να δράσουμε για την αξιοποίηση των κονδυλίων υπέρ των υποδομών. Τα τα κονδύλια μάλλον συνοχής, να αξιοποιηθούν για να υποστηρίξουμε αυτές τις περιοχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο και για τη χρηματοδότηση της Γεωργίας. Εδώ πιο πολύ εννοώ την ανάγκη να υπάρξει ανανέωση των ε, ποικιλιών που καλλιεργούνται στον τομέα της Γεωργίας και στα εσπεριδοειδή στο νότο της Μεσογείου. με ιδιαίτερα ε, κριτικό πνεύμα. Εδώ λοιπόν να επιφυλαχθώ για να σχολιάσω τα σημεία αυτά σε μια μελλοντική μου σύγηση. Ευχαριστώ πολύ μετά από όλες τις παρεμβάσεις, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε την προοπτική μιας γενικής συμφωνίας, ιδίως για τα θέματα των κλιματικών αλλαγών, για την απορρόφηση των κοντιλίων, για την απασχόληση των νέων. Να σας θυμίσω ότι έχετε στις 9 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, για να επιβάλλετε τις τροπολογίες σας, και να σας διαβεβαιώσω ότι σε ό,τι με αφορά την ουσία των σχολείων σας τη συμμερίζομαι και εγώ. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Λέιφ Ογκνάς της DG Radio και τον οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σχολιάσω καταρχάς την πρόοδο που έχει επιτελεστεί για το χρονικό διάστημα 14 έως 20 και να πω ότι υποκαθιστώ και τον Γενικό μου Διευθυντή, τον κύριο Λεμέτρα, και για σήμερα το απόγευμα. Μάλλον θα έρθει και εκείνο το απόγευμα, οπότε θα ακούσετε και τα δικά του σχόλια αργότερα. Σήμερα το πρωί τον αντικαθιστώ. Μερικέ παρατηρήσεις λοιπόν για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί εδώ. Τα νέα είναι θετικά. Έχουμε πρόοδο και έχουμε περάσει σε ταχύτητα κροαζιέρας όπως λέμε. Ιδίως μετά το 2015 και 2016. Και για να εξηγηθώ. Το ποσοστό επιλογής προγραμμάτων ε, είναι πολύ ψηλό. 83%. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη έχουν 83% των πληρωμών ε, ήδη για τα μελλοντικά προγράμματα. Βεβαίω υπάρχουν κάποιε πληρωμέ που πρέπει να ε, τι ε, εκτελέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό θα γίνει μελλοντικά. Για το ποσοστό επιλογή, λοιπόν, το ποσοστό που έχουμε τώρα είναι καλύτερο από αυτό που είχαμε από το 2007-2013. Είναι 2,5% παραπάνω για την ίδια περίοδο. 7-13. Εν είδη συμπεράσματο, λοιπόν, να πω ότι τα πράγματα πάνε καλά για την περίοδο 14-20 και περιμένουμε να υλοποιηθεί το 100% των προγραμμάτων στο το τέλος της περίοδου. Δύο ακόμα ζητήματα θέλω να θίξω. Πρόταση που περιλαμβάνεται στις τροπολογίες να αποκατασταθούν τα ποσά τα ποσά που είχαν μειωθεί από το Συμβούλιο Να ανασταλούν οι περικοπές λοιπόν και να ξαναδούμε την αρχική πρόταση της Επιτροπής όπως ζήτησε και η δική σας Επιτροπή. Merci beaucoup. Euh, j'aurais une question euh, complémentaire pour vous. Le... Ευχαριστώ μια ερώτηση προς εσάς. Το ποσοστό που αναφέρατε είναι κατά μέσο όρο ποσοστό Σωστά. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών και μεταξύ των διαφορών περιοχών τους. Υπάρχουν χαρακτηριστικά δείγματα ή κάποιες περιπτώσεις που δείχνουν ότι υπάρχουν αποκλίσεις. Να επιβεβαιώσω ότι βεβαίω είναι ο μέσο όρο αυτό για το ποσοστό και φυσικά υπάρχουν ε, διαφορετικέ επιδόσει μεταξύ των κρατομέλων και των περιοχών του. Όμω θα το αφήσω αυτό το σημείο προσχολιασμό για το απόγευμα, όταν θα συζητήσετε εκτενώ με τον κύριο Λεμέτρα και μπορεί να σα δώσει και πρόσθετε πληροφορίε. Σε κάθε περίπτωση είναι μέσο όρο το 83%. Ωραία. Θα το συζητήσουμε και με τον Γενικό Διευθυντή. Η παράκλησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εδώ είναι ήδη από τώρα να μας φέρει όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβή στοιχεία για να ξέρουμε τι συγκεκριμένα αποκλήσεις υπάρχουν μεταξύ κρατών και περιοχών και να δούμε εάν ταιριάζουν με τις κατηγορίες των περιοχών όπως έχουν οριστεί ή είναι απλώς ε, γεωγραφικές αποκλήσεις που ξεπερνούν τα όρια των κατηγοριών μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ε, εκ των προτέρων που θα στείλετε στη γραμματεία τα ακριβή δεδομένα. Να κλείσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό και να θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες ως τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα και θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία στις 2 και 3 Οκτωβρίου. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, ένα πολύ σημαντικό σημείο που αφορά τον κατεξιοσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού 1059-2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινή ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων που λέγονται και ΝΑΤΣ. Πρέπει να εξετάσουμε το σχέδιο αυτό κατά πράξη πράξης που επιφέρει τροπολογίες και αλλαγές ίσονος σημασία στα ΝΑΤΣ, στις ε, εδαφικές στατιστικές μονάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σχέδιο αυτό τροποποιεί παραρτήματα του κανονισμού για την ονοματολογία των ε, μονάδων, των στατιστικών μονάδων. Αυτό είναι μια ε, τακτική που επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια και σκοπό έχει να βεβαιώσει ότι οι εδαφικές στατιστικές μονάδες που χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανταποκρίνονται πλήρως στην ε, διοργάνωση που προβλέπουν και τα κράτη-μέλη τα ίδια. Στη Γαλλία, λόγω χάρη, είχαμε μια αλλαγή στις περιφέρειες, μια μεταρρύθμιση συνολικά. Ε, απαιτήθηκε μια σχετική προσαρμογή, αλλά και σε άλλες χώρες υπήρξαν τέτοιες αλλαγές. Η, ε, η προθεσμία για να καταλήξουμε σε ένα ε, ψήφισμα που θα περάσει και από την Ολομέλεια είναι η 8η Οκτωβρίου και με δυνατότητα παράτασης για δύο μήνες. Θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει το σχέδιο αυτό και το εξουσιόδο της και μετά θα δώσω το λόγο στους συντονιστές μας καθώς και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μιλέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την κατηγοριοποίηση των εδαφικών στατιστικών μονάδων ΝΑΤΣ είναι μια βασική άσκηση της στατιστικής. Χρησιμοποιούν μια τεράστια ποικιλία δεδομένων, θα το ξέρετε, τα ποσοστά ανεργίας, ο κίνδυνο φτώχειας, την ε, δυνατότητα σύνδεσης στο ευρυζωνικό διαδίκτυο και πάρα πολλά άλλα. Εδώ συλλέγουμε δείκτε για να αναλύσουμε τι οικονομικέ και κοινωνικέ επιδόσει των περιοχών, να δούμε ποιε έχουν πολύ καλέ επιδόσει, ποιε ε, καθυστερούν και να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε ημένα από του δε. Και βεβαίω που χρειάζεται πολιτική παρέμβαση. Ακολουθούμε τρει βασικέ αρχέ για τα ΝΑΤΣ, τρεις, ε, την σταθερότητα στον χρόνο, τη συγκρισιμότητα των περιοχών, και να τα αναλύσω. Η σταθερότητα στο χρόνο και η ε, διασύνδεση με τις εθνικές ανάγκες είναι δύο πράγματα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ε, διότι όταν αλλάζουν οι περιοχές ως προς τις επιδόσεις τους, χάνουμε την ιστορική πρόπτικη των πραγμάτων και κάποιες φορές χρειάζονται χρόνια για να τα αποκαταστήσουμε. Η σταθερότητα επίσης στη διάρκεια του χρόνου ε, επιβάλλει πολλές, ε, ε, πολλή δουλειά και κόπο από την πλευρά και τη δική μας της βάσης δεδομένων και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Πάντως, για τις υποδομές θέλουμε για όλες τις περιοχές να έχουμε στατιστικές, στατιστικά στοιχεία και αυτές που έχουν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα και αυτές που θα πάνε καλά. Αν υπάρχει όμω κατάλληλη διοικητική δομή στα κράτη-μέλη, συλλέγουμε πιο εύκολα τα δεδομένα και μπορούμε και πιο εύκολα να εφαρμόσουμε πολιτικά προγράμματα που μπορεί να πετούνται. Για τη συγκρισιμότητα των περιοχών, ε, κοιτάζουμε και τα όρια των, ε, ε, του αριθμού κατοίκων ανάλογα με, το, με τα κριτήρια που έχουμε ορίσει για τον ΝΑΤΣ, ώστε να διαχωρίζουμε σωστά μεταξύ ΝΑΤΣ e 2 και ΝΑΤΣ 3 που, ξεπερνάνε τους 8, που φτάνουν στους 8.000 κατοίκους ας πούμε ως περιοχές. Πάντως αυτό έχει να κάνει και με τη συγκεκριμένη περιοχή και το πώς ε, κατηγοριοποιεί και το κράτος μέλος στις διάφορες περιοχές. Πάντως ε, επιτρέπουμε και μια ε, κατά μέσο όρο απόκληση στον αριθμό των κατοίκων για τις αλλαγές των ΝΑΤΣ. Αναλόγως με το τι μας επισημαίνουν τα κράτη-μέλη, αλλάζουμε κατά τη διάρθρωση των περιοχών αυτών. Κάθε τρία χρόνια διοργανώνουμε μια επίσημη διαδικασία προσαρμογών και αλλαγών. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να μας κάνουν τις επίσημες προτάσεις τους και συζητούμε με ομάδες εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σε δημόσιες διαβουλεύσεις. Και μετά βεβαίω την έγκριση τη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Εντροπή, ερχόμαστε και εδώ. Αυτό που αλλάζουμε πάντως είναι απευθείας ε, το τι μας έχουν ζητήσει τα κράτη-μέλη. για τις αλλαγές λοιπόν, είχαμε μικρές αλλαγές σε πέντε χώρες μόνο, στο Βέλγιο, την Εστονία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στον Άτρια. Ε, κάποιες περιοχές άλλαξαν σύνορα στην ουσία, αλλά και στη Σαρδινία, στην Ιταλία και την Κροατία. Εκεί κάποιες περιοχές πέρασαν σε το επίπεδο ΝΑΤΣ 2. Αλλά είναι περιορισμένοι σε εμβέλειες αυτές οι φυλακές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Θα ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση με τους συντονιστές κατά πρώτον. Ο λόγος στον συνάδελφο Νόβακοφ για το ΕΛΚ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ξεκινάμε αυτή την πολιτική περίοδο με ένα τέτοιο θέμα. Προσπαθώ να βρω, αν θέλετε, ψυχή και πνεύμα σε αυτήν την δύσκολη και δυσανάγνωστη, θα έλεγα, στατιστική εργασία. Παρόλο που ακούσαμε ότι είναι ίσονος σημασίας και μάλλον τεχνικές, ε, κατά κάποιο τρόπο, αλλαγές, και ότι πρέπει να ανταποκριθούμε και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα κάποιων περιφερειών, είναι καλό να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές. Και σκεφτόμουν ότι ακριβώς επειδή κάποιες περιοχές βρίσκονται δίπλα σε κάποιες άλλες και καλύπτουν παρόμοιες ε, απαιτήσει και παρόμοια δεδομένα όσον αφορά παραδείγματος χάρη τον πληθυσμό, και την ίδια ώρα βλέπουμε ένα δήμο, μια κοινότητα να είναι καθαρά αγροτική και μια άλλη βιομηχανική ή με προσανατολισμό προς τον τουρισμό να πρέπει να εφαρμόσουν ίδιες προδιαγραφές και πολιτικές. Δεν ξέρω τι μαγική λύση θα βρούμε, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την κάθε κοινότητα, τον κάθε μικρό δήμο και να ανταποκριθούμε στις δικές τους απαιτήσει και προδιαγραφές. Παραδείγματος χάρη, ένα μικρό χωριό, μια μικρή κοινότητα που ακόμα δεν έχει, παραδείγματος χάρη, σύνδεση με το σύστημα υδροδότησης. Αυτό είναι η πολύ σημαντική απέτηση για τη συγκεκριμένη περιοχή και βεβαίως ε, με μεγάλη χαρά θα ακούσω την απάντηση της Επιτροπής όταν ε, και οι συνάδελφοι σχολιάσουν. Δεν ξέρω, έχετε λύσεις για κάτι τέτοιο. Πραγματικά αυτό θα είναι κάτι που σίγουρα θα ανταποκρίνονταν πολύ καλύτερα στις ανάγκες ε, όλων των περιοχών. Ευχαριστώ. Σκρέλα για τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα που όλοι ξεκουράστηκαν, ελπίζω όλοι να ξεκουράστηκαν μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και μπορούμε να ξαναρχίσουμε τη δουλειά μας και να προχωρήσουμε. Η έκθεση αυτή είναι μια τεχνική έκθεση και φυσικά ανταποκρίνεται στο κατά πόσο έχουν δώσει με επιμέλεια τα κράτη-μέλη τα στοιχεία που ανταποκρίνονται στις ε, μικρές διορθώσεις ε, που αφορούν τις περιφέρειες και τις ε, εδαφικές οριοθετήσεις. Δεν έχω συγκεκριμένα σχόλια να κάνω, αλλά αναφερθήκατε σε κάποιους δείκτες. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αναφέρθηκε σε κάποιους δείκτες. Μπορείτε να μας πούτε κατά πόσο το Brexit επηρεάζει, γιατί κάπως θα γίνει αυτό το Brexit με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πώς επηρεάζει αυτό εδώ το συγκεκριμένο θέμα. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον ε, όσον αφορά τους μέσους όρους που μας δώσατε και τις οικονομικές ε, επιδόσεις και τους δείκτες θα επηρεαστούν από το Brexit. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσετε την κατανομή και την κατηγοριοποίηση των περιφερειών θα ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα, θα τα προσαρμόσουμε στη νέα κατάσταση μετά το Brexit. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα υπάρξει στατιστική επίπτωση και αντίκτυπος. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Σας ευχαριστώ, Κωνσταντ. πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και θα περιμένουμε την απάντηση της Επιτροπής. Ο Αντρέη για τη Renew. Ευχαριστώ. Έχω μια διαδικαστική ερώτηση. Τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τα νέα στοιχεία και ζητούν ε, κάποιες προσαρμογές και αλλαγές. Αυτό δικαιολογείται, υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευσης, ανταλλαγής ε, πληροφοριών. Πώς ακριβώς γίνεται. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Νίκλας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίσατε όλοι. Ελπίζω να περάσετε όμορφες διακοπές. με μεγάλη χαρά αυτό που είπε ο κύριος Νόβακοπ. Όντως, η κάθε περιφέρεια έχει ειδικέ ανάγκες και θα πρέπει να υπάρξουν λύσεις που να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ειδικέ ανάγκες. Είναι θέμα κατηγοριοποίησης, αλλά όχι μόνο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι η αποκέντρωση, η αποκεντρωμένη προγραμματική οργάνωση είναι κάτι που σας έχει απασχολήσει και πώς σκέφτεστε να ανταποκριθείτε σε αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Για την ομάδα Ίντε, ο Αλεσάνδρο Μότσα. Όχι. Η κυρία Ντονάτο. Ε, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τα σχόλια των συναδέλφων. Ιδίω με τον συνάδελφο από τους πράσινου τον κύριο Νίνα, που μίλησε πριν από μένα. Είναι σημαντική η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εντοπισμό νέων εδαφικών στατιστικών μονάδων και επίσης σημαντικό είναι εκτός των στατιστικών δεδομένων και των παραδοσιακών δικτών να κοιτάξουμε και πτυχέ και διαστάσεις που μπορούν απευθείας να επισημάνουν οι συνεργάτες μας στις διάφορες ε, περιοχές επιτόπου. Αυτά πολλές φορές μπορούν να διαφεύγουν από τις συλλογές στοιχείων, από τις στατιστικές υπηρεσίες και μπορούν να είναι και ε, ιδίω ιδιαίτερο σημαντικά. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όποιο ασχοληθεί με τη νέα κατηγοριοποίηση ε, να ορίσει καλύτερα τις ανάγκες και το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης των διαφορών περιοχών Θα ήταν λοιπόν καλό και αυτές οι πτυχές να αναλυθούν σωστά και να δώσουμε το λόγο και στους επιτόπους συνεργάτες μας και εκπροσώπους μας στις περιοχές για να είναι ακόμα πιο πλήρη τα στοιχεία που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ομάδα μεταρρυθμιστών συντηρητικών ο Ραφαέλα Φίτο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις που μας έδωσε ήδη η Επιτροπή Θεωρώ ότι λίγα μπορεί να πει κανεί και να σχολιάσει και να συζητήσει όσον αφορά αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Μια ερώτηση να κάνω προς την Επιτροπή. Ωραία είναι αυτά που λέτε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις. Όμως, επί του περιεχομένου υπάρχουν κάποιες σημαδιακές και χαρακτηριστικές αλλαγές για κάποιες περιφέρειες. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτά τα νέα στοιχεία πώς μπορεί να επηρεάσουν κάποιες περιφέρειες θετικά ή αρνητικά. Εγώ νομίζω αυτό θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, Μαρτίνα, καταλάβαμε ότι εσύ εκπροσωπείς την GUE NGL και όχι το ECR. Και τώρα θα ακούσουμε τον Ραφαήλ από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές στην ECR ομάδα πολύ γρήγορα να πω ότι όπως δικαίως θύμισαν οι συνάδελφοι, πρόκειται για μια ε, αξιολόγηση, μια ε, προσαρμογή τεχνικού χαρακτήρα για να καταλάβουμε καλύτερα και πώς γίνονται οι δαπάνες, αλλά και τα τεράστια, τις τεράστιες δυσκολίες που εξηγούν τις ε, καθυστερήσεις και τις διαφορές, τι αποκλήσει, θα το δούμε. 3% ακούσαμε ότι είναι το ποσοστό απόκλησης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ε, τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή να δούμε κατά πόσον μπορεί να ορίσει τις ανάγκες ε, αλλαγών και προσαρμογών περιοχή ένα περιοχή. Είναι τεχνικά τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να καταλάβουμε πώς στην πραγματικότητα τα επιμέρους κατημέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ε, σόρευση και τον συνδυασμό με τα εθνικά κονδύλια για να αξιοποιήσουν ως το δυνατόν καλύτερα αυτά τα αυτούς τους Είναι λοιπόν τεχνικού χαρακτήρα ο κανονισμός και αλλαγή του, όμως θα έχει τεράστιο πολιτικό αντίκτυπο και ε, στην ανάπτυξη των ε, επιμέρους περιοχών. Σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς θα ήθελε το λόγο. Ο κύριος Ροπέ και μετά ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι οι τροπολογίες είναι τεχνικής φύσης και αφορούν μόνο τις πέντε χώρες που μας ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν όμως ο τρόπος που διαιρούνται οι περιφέρειες ε, στηρίζεται σε κριτήρια και ένα από αυτά είναι το ΕΠ. Και αυτό το κριτήριο χρησιμοποιείται ως βάση για τον προσδιορισμό των καλαθιών για την υποστήριξη των διαφόρων περιφερειών. Αυτό είναι όμως πολιτικό θέμα περισσότερο. Έχουμε κάποιες ε, διαφοροποίησεις γιατί μπορεί να έχουμε μια χώρα σε επίπεδου με φτωχές κάποιες από τις περιφέρειές της. Οπότε το ΑΕΠ δεν είναι επαρκές κριτήριο. Επίσης, δεν είναι πάντα οι ίδιες επιδόσεις των κρατών μελών και όλες οι πρωτοβουλίες δεν είναι εξίσου σωστές. Και μερικές φορές ο διαχωρισμός ε, των περιφερειών σε διάφορα επίπεδα στόχο έχει να μειώσει τις διαφορές μεταξύ τους. Μετά όμως ε, τα κράτη αποφασίζουν πώς θα, ε, που θα βάλουν τα σύνορα μεταξύ των διαφόρων ε, εδαφικών μονάδων στην επικράτειά τους. Θα πρέπει όμως, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει μεγάλες διαφορές εντός του ίδιου κράτους μέλους, να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες γιατί μερικές φορές είναι πολύ χρονοβόρες οι στατιστικές διαδικασίες. Το 2016 έγιναν κάποιες αλλαγές σε τέσσερις χώρες συμπεριλαμβανομένες και της δικής μου πατρίδας, της Λιθουανίας. Και δυστυχώς ε, για την περίοδο 2021-2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τα στοιχεία της με βάση την προηγούμενη νομοθεσία που ίσχυε του 2013 και όχι τη αλλαγή τη νομοθετική που έγινε το 2016. Για δύο όμω χώρε, την Πολωνία και τη Λιθουανία, εν προκειμένου, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να ζήσουμε βάσει τα στοιχεία όχι του 2016, τα νέα στοιχεία, αλλά του 2013. Ενώ είναι εμφανεί οι αλλαγέ που έχουν γίνει. Γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ε, νομοθετικές αλλαγές που έγιναν και να τις χρησιμοποιήσει στα έγγραφά της για τους κανόνες της συνοχής και τα χρηματοδοτικά της πακέτα. Η δεμή θα είναι ισμάτιν όλες οι αλλαγές που κάναμε. Και οι αλλαγές που γίνονται σήμερα θα ληφθούν υπόψη για την περίοδο μετά το 2034. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας ε, συγχρονισμός των αλλαγών με τα, τις, τα μέτρα που εφαρμόζονται. Ο κύριος Μπούντα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση είναι τεχνική μεν, αλλά πολύ σημαντική ιδέα γιατί αφορά την ανάπτυξη, τη δυνατότητα εκταμίευσης και απορρόφησης των ε, κοινοτικών κονδυλίων από τις περιφέρειες, τις μικροπεριφέρειες και άλλους φορείς. Και θα θέλαμε να συστήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την ε, δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλίων, περνώντας από κάποιες συνεταιριστικές ε, ή συνεργατικές δομές. Όταν υπάρχει μεταρρύθμιση που δίνει την ευκαιρία σε διάφορες ε, περιφέρειες ή δήμους να εκταμιεύσουν τα κονδύλια. Στη Δυτική Ρουμανία έχουμε τρεις δήμους της ίδιας περιφέρειας που συνεργάστηκαν για να εκταμιεύσουν περισσότερα κοινοτικά κονδύλια. Στη Ρουμανία πολύ συχνά ακούμε ε, τη μορφή ότι οι Βρυξέλλες δεν μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια. Θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία λοιπόν στις περιφέρειες αυτές να βελτιώσουν την ικανότητα απορρόφησής τους ακόμη και αν δεν είναι μέσα αναγνωρισμένε από την κυβέρνηση. Θα πρέπει τα κονδύλια να φτάσουν στι περιφέρειε ανάλογα με τι ανάγκε του. Και δεν θα πρέπει να κολλήσουμε, να μείνουμε κολλημένοι ε, σε κάποιε νομοθετικέ διατάξει. Δεύτερο ε, ζήτημα που με προβλημάτισε στη Ρουμανία είναι η ανάπτυξη των δικτύων υποδομών. Κυρίως ε, των υποδομών της ίδρευσης, ιδροδότησης. Κάποιες Κάποιοι δήμοι έχουν πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια κονδύλια. Αν λάβουμε όμω υπόψη την ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών, δεν μπορούμε στι Βρυξέλλε να ορίζουμε ποιε περιφέρειες θα δικαιούνται πρόσβαση στου πόρου και τα κονδύλια. Θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να λαμβάνονται αυτέ οι αποφάσει. Το κράτο να αποφασίσει ποιοι φορεί και ποιε περιφέρειες θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ενισχύσεις και όχι να γίνεται κεντρικά αυτός ο προσδιορισμός από τις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς παρακαλώ, θέλει το λόγο. Από ό,τι βλέπω, όχι. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι αυτή η στατιστική μεταρρύθμιση είναι ε, ίσονος σημασίας. Γιατί η πρόταση που μα υποβάλλατε δεν κατηγοριοποιεί τις περιφέρειες των κρατών μελών. Προσδιορίζει μόνο κάποια γεωγραφικά όρια των στατιστικών περιφερειών. Και είχαμε και άλλους κανονισμούς ΝΑΤΣ που ήταν πολύ πιο σημαντικοί μίζωνος σημασίας. Παρ' όλα αυτά, δίκιο έχετε ότι οποιαδήποτε στατιστική μεταρρύθμιση έχει και ένα πολιτικό αντίκτυπο. Και γι' αυτό έγιναν συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να μεριμνήσετε και να δώσετε απαντήσεις. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αυτές οι στατιστικές αλλαγές θα έχουν για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού επίπτωση στη κατανομή των κονδυλίων οι στατιστικές αυτές δηλαδή τροποποίησεις είναι τέτοιες εμβέλειας ώστε να επηρεάσουν την κατανομή των κονδυλίων ε, στις διάφορες χώρες και περιφέρειες. Έχετε το λόγο και παρακαλώ μην ξεχάσετε και την ερώτηση για το Brexit που έγινε, που επίσης είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπα, ρωτήσατε αν οι αλλαγές θα έχουν ε, επιπτώσεις στις, στα δημοσιονομικά κονδύλια. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Ε, στα τέλη του έτους θα εφαρμοστούν οι αλλαγές, αλλά τα στοιχεία για αυτές τις νέες στατιστικές μεταρρυθμίσεις θα αρχίσουν να έρχονται από τον Ιανουάριο του 2021, οπότε δεν μπορώ να προβλέψω ότι επιπτώσεις θα έχουν στα δημοσιονομικά κονδύλια. Ε, συνήθως ε, για τα δημοσιονομικά κονδύλια ε, καταρτίζουμε τριετή μέσου όρου. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι θα γίνει από το 2021 και μετά, πώ θα αναπτυχθούν οι περιφέρειε, τι χαρακτηριστικά θα έχουν. Νομίζω ότι γενικώ δεν θα υπάρξουν αλλαγέ, αλλά θα χρειαστούμε φυσικά χώρο για να, χρόνο για να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τι πληροφορίε και να απαντήσουμε πιο σχολαστικά. Και την ερώτηση αυτή καλύτερα να τη θέσετε στο Μάρκ Λεμέτρη, γιατί η Γενική Διεύθυνση ΡΕΓ είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά για το πώς αντιμετωπίζονται οι περιφέρειες με παρόμοια προβλήματα και αν εξετάζουμε τις μεμονωμένες ανάγκες των Δήμων και Περιφερειών και πώς μπορούμε να εστιάσουμε καλύτερα τις ε, δαπάνες, ώστε να έχουμε πιο στοχοθετημένες δαπάνες. Αυτή την ερώτηση καλύτερα να την θέσετε στον ε, Διευθυντή Λεμέτρ, γιατί εγώ είμαι περισσότερο αρμόδιος για τα τεχνικά θέματα του κανονισμού. Ε, ρωτήσατε για το Brexit. Ε, το σκεφτήκαμε και στα θέματα της ταξινόμησης του ΝΑΤΣ. Έχουμε οικονομικές, ε, οικονομικά εδάφη και προς το παρόν, πριν το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να το βγάλουμε από τώρα. Για το Brexit, ε, ίσως χρειαστεί ένας γενικός κανονισμός, omnibus, που θα τροποποιεί όλες τις ε, νομοθετικές πράξεις που θα χρειαστεί να αλλάξουν λόγω του Brexit. Πάντως, σε θέματα ΝΑΤΣ θα χρειαστούν παραρτήματα για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές σε περίπτωση που υλοποιηθεί το Brexit. Τώρα, τα αιτήματα των κρατών μελών, αν συμπεριλαμβάνονται. Από ό,τι ξέρω, ανέκαθεν ε, συμπεριλαμβάνουμε τις αλλαγές που ζητούν τα κράτη-μέλη στον κανονισμό ΝΑΤΣ. Εμείς κάνουμε ένα σύντομο έλεγχο για το αν ισχύουν οι, κανονι... διατάξεις του ΝΑΤΣ και είναι συμβατοί με τα αιτήματα, αλλά δεν απορρίπτουμε εμείς αιτήματα. Και υπάρχουν κάποιες παρεκκλήσεις, εξαιρέσεις λόγω περιβαλλοντικών, ιστορικών, πολιτιστικών ε, αιτίων. Αλλά από ό,τι ξέρω, ανέκαθεν να κάναμε δεκτές τις προτάσεις των κρατών μελών. Ενδιαφέρον ήταν το σχόλιο όχι μόνο να εξετάσουμε τους δείκτες στατιστικών στοιχείων, αλλά συγκεντρώνουμε πληροφορίες και από τον κόσμο επιτόπου. Ε, πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται κατά ανάγκη στα στατιστικά δεδομένα. Φυσικά κάνουμε και έρευνες, κάνουμε δημοσκοπήσεις ε, στις μεταφορικές εταιρείες, ε, στους δήμους και εκεί έχουμε άμεση επαφή με τον κόσμο. Συνήθως όταν έχουμε μια έρευνα, ρωτάμε τον κόσμο ποια είναι η θέση του για την παρούσα κατάσταση. Ρωτάμε αν είναι άνεργος ή όχι. Και επίση ε, με τα big data, τα μαζικά δεδομένα, με τα ανοιχτά δεδομένα έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Και φυσικά αν έχετε προτάσεις, πολύ ευχαρίστω να τις ακούσουμε για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τέτοια δεδομένα. Και κάτι άλλο Μας είπατε ότι είναι χρονοβόρες, χρονοβόρες οι διαδικασίες. Το ΝΑΤΣ 2016 δεν χρησιμοποιήθηκε ακόμη για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών προτάσεων για το επόμενο ΠΔΠ. Και στηριζόμαστε στο ΝΑΤΣ 2013, στην προηγούμενη εκδοχή του κανονισμού. Και όντω υπήρξαν αλλαγέ στη συνέχεια. Και η κατεξοδότηση πράξη παρόμοιε ήταν. Όντω είναι χρονοβόρε οι διαδικασίε. Το πρόβλημα όμω είναι ότι στο ΝΑΤΣ του 2016 είχαμε στοιχεία από την 1η Πρώτου 2018 και χρειαζόμαστε τριετής μέσους όρους για να υπολογίσουμε τις δημοσιονομικές προτάσεις. Έχουμε λάβει μερικά στοιχεία γιατί κάνουμε μια προσπάθεια τα κράτη-μέλη να μας δώσουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ, για την απασχόληση που είναι τα πιο σημαντικά που λαμβάνονται υπόψη στους ε, υπολογισμούς. Αλλά Τώρα αρχίζουμε με τον ΑΣ 2018 να δημιουργούμε το τριετές, τον μέσο όρο. Και χρειάζεται χρόνος γι' αυτό. Και τώρα τι περιφέρεις κάνουν κάτι τέτοιο και αυτά ρωτήσατε στον Μάρκ Λεμέτρ για να σας πει αν, έχουν αλλάξει, αν έχει αλλάξει τίποτα σχετικά. Yeah, that's, what I can say. It's Αυτά νομίζω μπορώ να πω προς το παρόν εκ μέρους της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις που μας δώσατε και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση μας έδειξε ότι δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει αντίρρηση για τον κανονισμό αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ότι η εξέταση του παρόντος κανονισμού μπορεί να προχωρήσει. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αναφέρθηκε στη συζήτηση που θα έχουμε με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Λεμέτρα, σήμερα το απόγευμα. Σας καλώ όλους να είστε παρόντες το απόγευμα. Είναι μια σημαντική συνάντηση, καθότι αναμένουμε τον νέο επίτροπο. Μπορούμε λοιπόν εν να συζητήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιφερειακών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. θα ακολουθήσει η συνεδρίαση των συντονιστών και καλώ όλους όσους δεν είναι συντονιστές και δεν συμμετέχουν στην συνεδρίαση αυτή να εγκαταλείψουν σιωπηλά και γρήγορα την αίθουσα. Στις 3 σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσουμε εκ νέου.